Ο Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου από δυο λόγια στην αρχή. Κατά τη διακοπή της Συνόδου μου επισημάθηκε ότι σήμερα στο Αφγανιστάν φωνεύτηκε Ιταλός στρατιώτης σε αυτή την ε, αποστολή που έχει διεξαγάγει το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Και ε, ξέρουμε ότι τον τελευταίο μήνα σκοτώθηκαν 15 Βρετανοί στρατιώτε. Οπότε να θυμόμαστε άντρε και γυναίκε οι οποίοι υπηρετούν σε ενόπλε δυνάμει. Οι οποίοι επιτελούν κάποιε αποστολέ στο εξωτερικό σε ιδιαίτερε ευγενεί συνθήκε. Επομένω, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν του ξεχνάμε. Και σα ευχαριστώ.